Στου στους ε, παραγωγούς για το σύστημα. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε τη συζήτηση καθώς και τη σημερινή Ολομέλεια. Η επόμενη θα λάβει χώρα αύριο 21 Απριλίου, ξέρετε, από τις 9 μέχρι 1 και 3 μέχρι 7 το βράδυ. Δηλαδή Αύριο θα λυθεί